2013. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης. Και θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην πρώτη μας σύνοδο της Ολομαλίας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ξεκινήσω δυστυχώς με μια δυσάρεστη ε, είδηση. Ο συνάδελφο Λόταρ Μπίτσκι ε, πέθανε απρόσμενα στι 13 Αυγούστου. Ο ξαφνικό του θάνατο ε, μα έπληξε όλου όλοι τον εκτιμούσαμε ιδιαίτερα ε, και έχερε ε, εκτίμηση από όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, χάσαμε έναν πολιτικό, ο οποίος ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομάδας της Αριστεράς άφησε το στίγμα του και στην Γερμανία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Χάσαμε έναν ειλικρινή φίλο ήταν ένας ιδιαίτερα μορφωμένος και ικανός συνομιλητής και θα τον έχουμε πάντοτε στη μνήμη μας με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο θάνατος του Λότερ Μπίτσκι είναι σοβαρή απώλεια για το Κοινοβούλιο και είναι μια οδυνηρή απώλεια για την οικογένεια και για τους φίλους του. Η σκέψη μας είναι κοντά στους δικούς του ανθρώπους και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κρατήσουμε ένα λεπτό σιγής. Ευχαριστώ.